in June, uh, where the parliamentary scrutiny will be discussed, the, the rule of law and the role of national parliaments in uh, protecting... Ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων για την προστασία του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι θέμα της συζήτησης και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και μετά ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το Ελληνικό Συνέδριο και βέβαια Άσταση με τα μεγαλύτερα θέματα μάλιστα. Σημείο 3 στην ημερησία Σημείο 4. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων και θέλω να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Το μικρόφωνο της Πρόεδρου έχει κλείσει. Το μικρόφωνο της Πρόεδρου είναι κλειστό. Το μικρόφωνο της Προέδρου είναι κλειστό. Σήμερα δεν είναι. Γιατί είναι το μικρόφωνο μου, δεν κλείνω. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη έγκριση πρακτικών 19 Νοεμβρίου 3 Δεκεμβρίου στη διάθεση. αυτό uh, το τέλος συνεδριάσεως ε, δεν γερθούν αντιρρήσεις, θα εγκριθούν και περνώ στο θέμα, το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δύο οργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία, έκθεση προετοιμασία ολομέλειας με τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεματικών, με την πρόεδρο της Επιτροπής Θεματικών Υποθέσεων για μια καλύτερη νομοθεσία, διοργανική συμφωνία που έχει υπογράψει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας ενημερώσω πως για την έκθεση αυτή έχουν κατευθεί 97 τροπολογίες. Ομιλώ για την έκθεση Χιούμπνερ για την ε, καλύτερη νομοθεσία. Τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί εγκαίρως. Για το 15 επίσης, το 15 έχουμε σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία που ήδη έχουν παληθεύσει οι, νομομαθείς, οι γλωσσομαθείς νομικοί και δικηγόροι έχει επαληθευτεί λοιπόν από τους γλωσσομαθείς δικηγόρους των τριών θεσμικών οργάνων και προσαρτάται στα, ε, στην έκθεσή μας εν ώψη της Ολομέλειας. All aspects of the interinstitutional agreement, so they cover the impact assessment. Καλέ, καλύπτουν ε, τις συνέπειες, την αξιολόγηση συνεπειών, το κανονιστικό υπερθεματισμό, τα την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου, Εθνικά Κοινοβούλια. Τροπολογίες έχουν καταθεί επίσης που σχετίζονται με το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου. Δεν καλύπτονται όμως από τη διοργανική συμφωνία στο συγγνώμη, διότι ορισμένε από τις τροπολογίες δεν καλύπτουν θέματα της διοργανικής συμφωνίας που αποτελούν προνομία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τα άλλα θεσμικά όργανα τις επιλογές μας. Θα βεβαιώ δε ότι προσπαθώ να δεχθώ στα δυνατόν περισσότερες ε, προτάσεις και να ενσωματώσω στα δυνατόν περισσότερες τροπολογίες στις συμβαστικές. Κάποιες από αυτές βεβαίως ήταν αντιφατικές μεταξύ τους. Και επίσης θέλω να επισημάνω πως έμφαση δόθηκε τις συνέπειες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εισαγωγή νέας νομοθεσίας. Άχθος, όπως είπαμε, επισκόπηση του άχθους, ε, και άλλα σχετικά θέματα. Σας διαβεβαιώ ότι γνώμονας μου για τις τροπολογίες ήταν μια θετική και επικοδομητική προσέγγιση των τροπολογιών ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση και με τους κοιόδης καταφέραμε ύστερα από μια συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου να καταλήξουμε σε πέντε συμβαστικές πρώτα και δύο ακόμη στη συνέχεια που ελπίζω ότι θα σας βρουν σύμφωνος. Αυτά έχω εγώ να σας πω. Και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση με τη συζήτηση για τις τροπολογίες, για την έκθεση, οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί σε σχέση με την έκθεση αυτή και έχετε το λόγο. Κύριε Στροχόφιστο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω ε, μία νέα συμβαστική τροπολογία F εάν είναι δυνατόν. Παράγραφος 12. 3β. Ε, εκεί που λέει ongoing discussion. Λοιπόν, μετά από συζήτηση με πολλούς συναδέλφους προτείνω ε, συμβιβαστική τροπολογία F επί της 12 ε, και αντί της τροπολογίας 86 να έχουμε το ακόλουθο κείμενο. Μπορώ να το διαβάσω αν μου δίνετε τη δυνατότητα. Λαμβάνοντα υπόψη τις, ε, τους όρους της συμφωνίας, το Κοινοβούλιο προσδοκά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τις προτάσεις της που θα καθορίζουν στόχους ε, ε, που ε, θα είναι συγκεκριμένοι όσον αφορά την μείωση του ελλείμματος στο τομείς ενώ ταυτοχρόνως θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των νομοθετικών στόχων. Πρέπει να σας πω ότι εμπνευστήκαμε από ένα αντίστοιχο κείμενο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ή ίσως αυτοί αντέγραψαν εμάς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Μπορώ να σας το δώσω κιόλα γραπτά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κατάφερα να το γράψω έτσι όπως το διαβάσατε, αλλά παρόλα αυτά καλύτερα να μας το δώσετε. Κύριε Μακιντάιρ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, η μεταρρύθμιση είναι μια διαδικασία η οποία δεν ε, σταματάει και ε, μάλιστα και στην επισκόπηση αναφέρεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκίφερ Χόφστατ για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι στην πρώτη σελίδα της επισκόπησης αναφέρεται ότι η νομοθεσία θα πρέπει να αποφεύγει υπερβολικό διοικητικό άχθος κυρίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη κατά κάποιο τρόπο από εκεί ξεκινήσαμε εμείς στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει έτσι ώστε να μειώσουμε τα, το ρυθμιστικό και ε, ε, λοιπό άχθος. Οπωσδήποτε μπορώ να ε, συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Φερχόφστατ για μια νέα συμβιβαστική τροπολογία F όπου μπορούμε ρητά να αναφέρουμε ότι προσδοκούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ε, οι οποίες θα καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση του άχθους σε σημαντικούς τομείς. Γιατί άλλωστε αυτό απορρέει και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και θα ήθελα να προτείνω και μία αιτιολογική αναφορά παραπάνω στην έκθεση την οποία συζητούμε τώρα που θα λέει ότι ε, σε σχέση με τα συμπεράσματα ε, της, της ε, συνεδρίας του Συμβουλίου της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου Τώρα ας αφήσουμε στην άκρη το ποιος είχε την ιδέα πρώτος αλλά ε, και να ε, ασχοληθούμε πραγματικά με τους στόχους και με την μείωση του βάρους γιατί αυτό είναι κάτι ιδιαίτερος προσφυλές σε εμάς και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με χαρά βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει και θα θέλαμε αυτό να το αναγνωρίσουμε μέσω μιας αιτιολογικής αναφοράς. Επίσης, ε, ε, στο IIA αναφέρεται ε, και το, αναφέρονται και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και νομίζω ότι αυτή η ιδέα της ετήσιας επισκόπησης άχθους είναι κάτι ενδιαφέρον και σημαντικό και αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, γιατί κάπου λέει ότι ε, θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική νομοθεσία, νομοθέτηση, καθώς επίσης ε, και ε, το επιπλέον ε, άχθος. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε απολύτως δεσμευμένοι όσον αφορά τον κοινό στόχο της μείωσης του άχθους στις διαπραγματεύσεις ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρωθυπουργό βεβαίω ήθελε και ειδική συμφωνία, αλλά στην ουσία αυτό που ήθελε και θέλει είναι να βελτιωθεί η κατάσταση για όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδεοδό ε, δηλαδή ε, μια μεταρρύθμιση η οποία θα λάβει χώρα με διαρκή τρόπο έτσι ώστε να βελτιωθεί ο τρόπο νομοθέτηση και νομίζω ότι κατά αυτή την ε, ε, άποψη όλη αυτή η συζήτηση είναι σημαντική βεβαίω για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντική και για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, εγώ μπορώ να συμφωνήσω απολύτω με, με τον νέο συμβιβασμό ε, και θα ήθελα να προτείνω να προσθεθεί και αυτή η νέα αιτιολογική αναφορά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακιντάιρ. Ελπίζουμε ότι θα στρίξετε και τις άλλες συμβαστικές προτάσεις αύριο στην ψηφοφορία. Ναι, έχουμε συνεργαστεί για τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπόρεσα να είμαι στους σκιώδεις εισηγητές ε, δυστυχώς. Ε, ναι, ξέρω ότι αντεκαταστάθηκα επάξια και είχα και τους συμβούλους. Ξέρω ότι λάβατε υπόψη σας μου την συμβιβαστική, οπότε ναι, τη στηρίζω. Ευχαριστούμε. Ρίτσαρτ. Όλοι θέλουμε να λειτουργεί η καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο κ. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα το πετύχουμε αυτό. Αυτή λοιπόν η διοργανική συμφωνία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι όμως μια διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθέτηση και όχι απλώς για να αποφεύγουμε τον νομοθετικό υπερθεματισμό, γιατί ορισμένοι δείχνουν να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτές γίνονται για κάποιο λόγο και γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη πλειοψηφία ενισχυμένη δική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Άρα τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και φτάνουμε εκεί. Και όταν το κάνουμε έχουμε ενιαίους κανόνες και όχι 28 διαφορετικούς κανόνες και αντιθετικούς μερικές φορές μεταξύ τους, άρα μειώνεται και το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεπώς η δικιά μου προσέγγιση της ε, ομάδας μου για την έκθεση και για τις συμβαστικές τροπολογίες είναι ναι, βεβαίως να αναφερόμαστε στο νομοθετικό υπερθεματισμό εφόσον όμως δεν ξεχνάμε και το στόχο της ε, εκάστοτε νομοθετικής ρύθμισης. Πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε και το κόστος της μη νομοθετικής ρύθμισης. Τι οικονομικό βάρος είναι αυτό για τους καταναλωτές, τι σημαίνει αυτό για την προστασία του περιβάλλοντος, τι σημαίνει για τους φορολογούμενους, τι σημαίνει για τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, άρα να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Τώρα έχοντας κοιτάξει τις συμβαστικές τροπολογίες, νομίζω ότι όντως υπάρχουν πράγματι κάποιες ε, διατυπώσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στις επιθυμίες μας. Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν ίσως περισσότερα πράγματα να μπουν ε, μέσα, αλλά για την ομάδα μου πιστεύω ότι εντάξει θα τις δεχτούμε. Επίσης, σημαντικό είναι, όπως ήδη ακούσαμε, η εκτίμηση αντικτύπου και η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου να λογοδοτεί στις πολιτικές αρχές, να μην τις αντικαθιστά, να μην τις παρακάμπτει. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή κατά τη γνώμη μου. Συνεπώς με αυτές τις ανησυχίες που όμως καθησυχάζονται πιστεύω σε αυτό το κείμενο μπορούμε να δεχτούμε τις συμβαστικές σας προτάσεις. Ευχαριστούμε Ρίτσαρντ, λέει Άλλος κανείς. Γκί Φερχόφσταθ, εκ μέρους της Άλντε. Γιατί μιλήσαμε για τις συμβαστικές προτάσεις, αλλά τι λέτε, η γενική στάση ποια θα είναι. Εγώ μιλάω, λέει ο κ. Φερχόφσταθ, και εκ μέρους της Άλντε. Οπότε ισχύει αυτό και για την πρόταση Μάκιντος για μια επιπλέον ε, αιτιολογική σκέψη, μια πρόταση που να αναφέρεται στη σοφία του Συμβουλίου. Για αυτή την περίπτωση, ε, δεν λέω ότι ισχύει πάντα. Για μια φορά συμφωνώ. Ο Κίφερ Χόφστατ όταν έφυγε από το Συμβούλιο φοβήθηκε ότι έφυγε και όλη η Σοφία από το Συμβούλιο μαζί. Ναι, αλλά τώρα αυτές τις μέρες φαίνεται ότι επανήλθε κάπως, λέει ο κ. Φερχόφστατ, στο Συμβούλιο η Σοφία. Πρόεδρος, καλώς. Άλλη πολιτική ομάδα. Όχι, δεν βλέπω. Νομίζω ότι δουλέψαμε σκληρά για τις συμβαστικές τροπολογίες μέχρι και πριν από λίγα λεπτά ακόμα. Έχει γίνει λοιπόν η δουλειά, οπότε αύριο ελπίζω να έρθουν να ψηφίσουν πρώτα πολλοί άνθρωποι, γιατί υπάρχουν και άλλες συνεδριάσεις, και ΑΦΕΤ και ΕΚΟΝ και άλλες συγχρόνως συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα. Είναι σημαντικό όμως να είναι εδώ οι συνάδελφοι για να ψηφίσουμε. Τίποτα άλλο. Ωραία. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την έκθεση αυτή, συνεχίζουμε. Στην έκθεσή σου, Γιώργη, 20 λεπτά. Θες τώρα να πάρεις το λόγο. Ναι. Μεγάλη χαρά και κατάπληξη αισθάνομαι που έχουμε χρόνο για το θέμα αυτό. Να σας πω δύο λόγια για το ιστορικό του. Υπάρχει ένα ψήφισμα από το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα μηχανισμό για το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Έκθεση ΛΥΜΠΕ. Η Σοφία Νετφέλτος, εσύ και θα έρθει αργότερα να μα μιλήσει. Πολύ χρήσιμο ήταν η μέθοδος της εργασίας που επέλεξε. Ε, συγκάλεσε όλους τους σκιώδεις, της ΛΥΜΠΕ και γενική πάντα και εμένα να συμμετάσχουμε σε εργασίες. Ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα εργασίας, ένα έγγραφο εργασίας, στην ουσία 8 έγγραφα εργασίας, όλοι μας. Εγώ ανέλαβα το κομμάτι που είχε το ρόλο για των ετησίων ε, συνεδριάσεων των κοινοβουλίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι στη διάθεσή σας. Και στη συνέχεια, μια εβδομάδα περίπου πριν, συζητήσαμε αυτά τα έγγραφα σε μια άλλη συνεδρίαση. Αυτή είναι η κατάσταση. Αναλαμβάνω εγώ τη γνωμοδότηση, η οποία βέβαια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ψηφοφορία, από την ορίσετε για την έκθεση της Σοφή, από την ορίση λίμπε. Ε, από την ε, συνεδρίαση αυτό που αποκομίζω είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κοινή αντιμετώπιση και νοοτροπία αντί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ε, όλα τα κράτη-μέλη και στα 28. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές να ισχύουν και στα 28 κράτη χωρίς εξαίρεση. Η ιδέα ενός συμφώνου που θα προσπρογράψουν όλα τα κράτη-μέλη έχει μάλλον πολιτικό χαρακτήρα ένα τέτοιο σύμφωνο φαντάζομαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μπορεί να συζητηθεί βεβαίω, αλλά και κάτι ακόμη κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται κοινό τόπο, αλλά πάλι δεν είμαστε και φιλεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, δύο διαδικασίες επί παραβά... έχουμε τη διαδικασία επί και το άρθρο 7. Και αν κανεί κάνει τον κόπο να διαβάσει το άρθρο 7, θα διαπιστώσει ότι και τι περιγράφεται ω πυρηνικό όπλο, ε, ουσιαστικά είναι άχρηστο. Άρα χρειάζεται ένα ενδιάμεσο όργανο μεταξύ της, ή μια ενδιάμεση διαδικασία καλύτερα μεταξύ διαδικασίας επί παραβάση και το άρθρο 7 η οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από κάποια νομική βάση. Άρα, εάν χρειαστεί και μόνο βέβαια με αλλαγή συνθήκες μπορεί να ε, θεσπιστεί μια νομική βάση για την ενδιάμεση αυτή φάση. Αυτά είναι τα κύρια σημεία για μένα, για το έγγραφο. Για τη δική μας επιτροπή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπησέλθω σε πολλές λεπτομέρειες όπως τις προοπτικές, ε, την προοπτική μάλλον της ΑΦΚΟ για τα θέματα αυτά. Φυσικά μας ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα της κυβέρνησης. Νομιμότητα κράτος δικαίου πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κρατικές, τι εθνικές αρμοδιότητες, πολύ πεδίο για συζήτηση. Επίσης, ήδη έχουμε αντιμετωπίσει, θέλω να επισημάνω, προτάσεις για κανονισμούς και θα πρέπει πιστεύω να εστιαστούμε περισσότερο στα συστημικά προβλήματα, το συστημικό κίνδυνο δηλαδή για, που προκύπτει από τις παραβάσεις των δικαιωμάτων. Επί τη βάση αυτών, θα καταγράψω και την ε, ογνωμοδότησή μου όταν ήρθε θα θα δώσω στο διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, ενδεχομένω δε και αντιπροσωπεία τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, δεν ξέρω ποιου άλλου ενδιαφερόμενου φορεί, εμπλεκόμενου φορεί με κυβερνητικέ οργανώσει. Και πρέπει να αποτελέσει αυτό μια όλο εξελισσόμενη διαδικασία, αν και δεν βλέπω να υπάρχει η για γραμματεία. Ο στόχος πάντως θα είναι να διευκρινίζονται πρακτικές ορισμοί της νομιμότητας του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία το σύμφωνο της Σοφίνετ Φέλτ πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Για μένα αυτό θα ήταν το ιδεώδες και τι δεν βλέπω να υλοποιείται από την μια μέρα στην άλλη. Εάν όμως εγκαθιδρυθεί αυτή η αντίληψη, η κουλτούρα θα λέγαμε του κράτους δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όμως ότι πρόκειται να γίνει από τη μέρα στην άλλη, δεν είναι διακόπτης ε, να, να δει και να σβήνει. Πρέπει όμως όλα τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν στις ίδιες έννοιες ε, και του ίδιους ορισμούς τα κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ταυτόχρονα με αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των ε, νομικών παραδόσεων πολύ απλά, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, δεν χρειάζεται, θα αναφέρω το παράδειγμα του ρωμαϊκού και του αγγλοσαξονικού συστήματος και του μείγματο αυτών που βρίσκεται, βρίσκουμε στην ε, Σκοτία. Όλα όμως αυτά νομίζω αποτελούν μία βάση. Όλα αυτά αποτελούν μία βάση της έκθεσης που θα προχωρήσει και όταν έρθει η ώρα περιμένω να ακούσω τις δικές σας προσθήκες. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι προετοιμάζει ο Τζόρτζ την γνωμοδότηση ε, και ε, σκέφτηκε να κάνει αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο αποτελεί καλή προετοιμασία για την γνωμοδότηση και είναι πολύ καλή ε, πρωτοβουλία. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, έχει κανείς την αίσθηση ότι η συζήτηση είναι πιο γενική, πιο ε, διαφανής, πιο σωστή. Δεν ξέρω αν κάποιος ε, θέλει να προσθέσει κάτι, να σχολιάσει κάτι σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Ο Ρίτσαρτ Νέβη όχι, τα κατάλαβε όλα. Τώρα, στις 4.30 έχουμε την ακρόαση και εκεί που είχαμε τόσα πολλά πράγματα και στην με μέση αδιάταξη, ξαφνικά έχουμε πολύ χρόνο. Νομίζω λοιπόν να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Okay, I, I still would, uh, yeah, would like to make today the presentation of the of what we decided at. Θα ήθελα να πούμε και να παρουσιάσουμε τα όσα ε, συνέβησαν και όσα ελέγχθησαν στην συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά καλύτερα να είναι περισσότεροι εδώ να έρθετε καλύτερα στι 4 και 20 αντί για τι 4.30 για να προλάβω να σα πω τα αποτελέσματα τη συζήτηση με του συντονιστέ.